Συνάδελφοι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Περιμένουμε. Γιατί το πρώτο θέμα που έχουμε μπροστά μας είναι η γνωμοδότηση της ΣΥΝΚΟ και ο εισηγητής δεν είναι μαζί μας ακόμα. Ξεκινάμε λοιπόν πάλι, λέει η Πρόεδρος. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. έγιναν προτάσεις για την τροποποίηση του 4 και 5, γιατί η συγγήτρια του πρώτου θέματος δεν είναι μαζί μας, οπότε μπορούμε να αλλάξουμε και να ξεκινήσουμε με το 5 για, την, για το διαφορετικό θέμα το οποίο προβλεπόταν εκεί. Καλώς λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι οι ανακοινώσει της Προέδρου. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο το οποίο θα ήθελα να θέσω. Και γι' αυτό συνεχίζουμε με ταχύτητα προώθηση της ισότητας και στα πλαίσια της ψυχικής υγείας. Η κυρία Μπεσέρα είναι η συγγήτρια. Έχουν γίνει στο παρελθόν αρκετές συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό. Έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες, αυτό δείχνει το επίπεδο ενδιαφέροντος και γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπεθέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και για τους συναδέλφους οι οποίοι όχι απλά ενδιαφέρθηκαν για το περιεχόμενο της πρότασής μου αλλά κατέθεσαν και αρκετές τροπολογίες οι οποίες βελτίωσαν νομίζω με σημαντικό τρόπο την ποιότητα θα ήθελα ίσως να αναφερθώ εδώ και στην εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε με τους Κιώδης από την πρώτη στιγμή, ιδιαίτερα σε σχέση με τις προτεραιότητες ε, τις οποίες έπρεπε να ορίσουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στην έκθεση. Και έχουμε συνυπογράψει αρκετές τροπολογίες, εγώ σαν εισηγήτρια και οι σκιώδεις συνεισηγητές μου. Διευκρινίζουμε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο την αρχιτεκτονική της έκθεσης αυτής. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταγγείλουμε μέσα από τα μέσα τα οποία προτείνουμε κάποιους μύθους και κάποια άλοθη τα οποία έχουν μέχρι τώρα χρησιμοποιηθεί γύρω από το θέμα αυτό. Έχουμε καταλήξει σε προτάσεις συμβιβαστικών τροπολογιών να γίνει στις 29 Νοεμβρίου η ψηφοφορία εδώ και τον Ιανουάριο η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Σε αυτή τη φάση Ε, θα έλεγα έχουμε φτάσει σε μια φάση όπου θα συζητήσουμε ακριβώς τη σχέση της γυναίκας και με την επιστήμη και με αυτού του είδους της ε, ε, καινοτομίες, την βελτίωση στον τομέα της έρευνας και την καινοτομία μέσα από την ισότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει μόνο έτσι ώστε να δοθεί ένας καινοτομικός χαρακτήρας που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τους μύθους και τις προκαταλήψεις αλλά να αποδείξουμε ότι και σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε σε θέση να κινητοποιήσουμε κάποιους μηχανισμούς τους οποίους έχει πάρα πολύ ανάγκη η κατάσταση των γυναικών σήμερα. Αύριο θα είναι πολλοί μαζί μας οι οποίοι έχουν προτάσεις γύρω από τις, από τα, τις προτάσεις και τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα. Αύριο θα συζητήσουμε ειδικότερα σημεία και για τη σχέση γυναικών και υγείας. Να πω ότι η έκθεσή μου ελπίζω πριν από οτιδήποτε άλλο να είναι χρήσιμη, τίποτα άλλο προς το παρόν. Ευχαριστώ κυρία Βεσέρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θα ήθελαν το λόγο. Θα ήθελα να καλωσορίσω ένα νέο μέλος στην Επιτροπή μας. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία μαζί του. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε προς το κοινό καλό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για, τις, ε, για τα καλά σας λόγια. Εγώ αντικαθιστώ το Σεμπαστιά. που είναι σκιώδης ε, εισηγητής, ε, ένας από τους σκιώδης ε, για την γνωμοδότηση και άλλων επιτροπών. Να πω ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το κείμενο και από την πρόταση της εισηγήτριας ελπίζει ότι η Επιτροπή Γυναικών θα μπορέσει να ενσωματώσει κάποια από τα στοιχεία τα οποία προτείνει η Επιτροπή Ανάπτυξης, Ανάπτυξης έτσι ώστε να ενισχυθούν τα εθνικά συστήματα υγείας και να υπάρξει ένα καθολικό σύστημα προστασίας της υγείας των πολιτών και να ζητήσουμε από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν κάνουν τις λεγόμενες μαζικής κλίμακας κλινικές δοκιμές Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να καλύψουμε και τις ανάγκες κατηγοριών εύθραυστων της κοινωνίας όπως και τις γυναίκες. Να δούμε επίσης τι γίνεται και στις φτωχές χώρες όπου η κοινωνική προστασία πρέπει να ενισχυθεί κατά πολύ. Νομίζω ότι αυτές είναι οι βασικές ιδέες που διακρίνουν την έκθεσή σας και θα τις λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα πριν από λίγο σκεφτόμουν την ιστορία των γυναικών και την ιστορία των ε, ψυχικών ασθενειών που πλήττουν τις γυναίκες. Πολλά χρόνια πριν εργαζόμουν σε ένα ίδρυμα για άτομα που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Υπήρχαν πολλές γυναίκες εκεί σε αυτό το Ίδρυμα, το, οι οποίες γυναίκες τώρα πολλές φορές θα πίστευε κανείς, μάλλον θα έλεγε κανείς ότι, θε, ότι έχουν άλλε, άλλου τύπου ασθένειες. Υπήρχαν μάλιστα κάποιες ε, μέθοδοι περίθαλψης των γυναικών που ε, θεωρούνταν μαγκανίες, μαγείες, με βότανα κτλ. Πρέπει λοιπόν να δούμε τη διάσταση του φύλου, να δούμε την πολιτισμική διάσταση, η οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Υπάρχουν μάλιστα ε, πολλοί που πίστευαν πως η μήτρα μιας γυναίκα δεν είναι σταθερή σε ένα σημείο, αλλά περιπλανάται στο σώμα της. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες αντιλήψει οι οποίες πρέπει να αλλάξουν. Και συμφωνώ με την ε, Μπέατρη ε, για αυτά που πρέπει να γίνουν και θα ήθελα να την ευχαριστήσω καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Χάρηκα πολύ που κατάφερα να συνεργαστώ μαζί τους. μπορέσαμε μαζί να συνυπογράψουμε πολλές τροπολογίες και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία. Πιστεύω πως οι τροπολογίες μας έχουν οδηγήσει σε ένα πολύ καλά δομημένο κείμενο που πιστεύω θα συνεισφέρει στην βελτίωση της ψυχικής υγείας των γυναικών στις κλινικές δοκιμές φαρμάκων γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε το ρόλο των γυναικών ε, στην κοινωνία και να δούμε την ε, διάσταση της υγείας, ψυχικής και σωματικής. Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία που θα συμπεριλαμβάνει και τη διάσταση του φύλου. Χρειάζεται να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση η οποία θα φορά όλο τον κύκλο ζωής ενός ανθρώπου από τη γέννησή του μέχρι τα γυρατιά. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη διάφορες ευάλωτες ομάδες, οι γυναίκες πρόσφυγες, ΛΟΑΔ και να πω ότι αυτά είναι θέματα με τα οποία ήδη ασχολούμαστε στην Επιτροπή αυτή. Μάλιστα είχαμε και ένα ψήφισμα για την Παγκόσμια ημέρα της ε, γυναίκας που αφορούσε τις γυναίκες πρόσφυγες. Χρειάζεται όμω να πιέσουμε για να γίνουν περισσότερες ε, δράσεις για τα κορίτσια και για τα αγόρια, για τα παιδιά, τα οποία υποφέρουν από διάφορα στερεότυπα σχετικά με το φύλλο. Χρειάζεται λοιπόν μία στρατηγική ισχυρή για την ψυχική υγεία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική και επίγουσα. Και θα ήθελα να στείλω αυτό το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και να... Ε, πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις κλινικές δοκιμές πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες ενέργειες, να συμπεριληφθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς έτσι ώστε να ε, συμπεριλαμβάνονται οι γυναίκες ως ε, ε, συμμετέχουσες σε διάφορες κλινικές δοκιμές γιατί πολλές φορές τους χορηγούνται φάρμακα τα οποία δεν ταιριάζουν σε αυτές. Είναι φάρμακα τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί σε γυναίκες. διάφορες θεραπείες οι οποίες δεν χρησιμεύουν σε τίποτα, δεν λύνουν το πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των γυναικών, όλων των γυναικών, ακόμα και των γυναικών εδώ σε αυτή την αίθουσα. Γι' αυτό λοιπόν είναι καθήκον μας να αναλάβουμε δράση. Θέλω λοιπόν να πω εδώ ότι θα καλωσορίσουμε κάθε συνεισφορά από όλες τις πολιτικές ομάδες και θα συνεργαστούμε με τους κοιόδης έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα συνεκτικό και πλήρες κείμενο. Θα σας δω λοιπόν πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ward. Κυρία Πετήρη, Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ πως η έκθεση είναι πολύ σημαντική, γιατί καλύπτει τις κλινικές έρευνες και την ψυχική υγεία. Υπάρχουν όμως ορισμένα προβληματικά σημεία. Στην πρώτη τη λογική σκέψη, ας πούμε, αναφέρεται ότι το δικαίωμα στην υγεία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα όμως εδώ υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Ε, αυτό το άρθρο δεν αναφέρει κάτι τέτοιο αναφέρει αντίθετα ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ίση πρόσβαση σε ε, περίθαλψη σύμφωνα με τις ε, προϋποθέσεις και των διεθνών διατάξεων. Το δικαίωμα στην ψυχική υγεία είναι δικαίωμα στη ζωή. Ωστόσο, δεν γίνεται σεβαστό το άρθρο αυτό στην έκθεση. Δεν ε, είναι σωστή η παράθεση. Επίσης, αναφέρεται το δικαίωμα στην άμβλωση. και επίσης το δικαίωμα της, ε, της ενσυνείδητης αντίρρησης. Όλα αυτά ανοίγουν στα θεμελιώδη λοιπόν δικαιώματα. Και πρέπει να δούμε, να δούμε μάλλον ότι εδώ υιοθετείται μια πιο ιδεολογική προσέγγιση παρά πρακτική κάτι που δεν βοηθά τις γυναίκες στην ουσία. ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ την ε, εισηγήτρια. Έχουμε ξανασυζητήσει αυτή την έκθεση στο παρελθόν και όπως και οι συνάδελφοι έχω καταθέσει τροπολογίες. Όπως και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση, διότι τονίζουμε πόσο σημαντική είναι η ψυχική υγεία όλων των γυναικών και αντιμετωπίζουμε τα θέματα των σχετικών παθήσεων καθώς ε, και τις, ε, τα συνδέουμε, το συνδέουμε αυτό το ζήτημα με τις κλινικές δοκιμές ε, και τη, τα όσα συζητούμε για τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Θέλουμε φυσικά να επιτύχουμε μεγαλύτερη ισορροπία και ισότητα για την πρόσβαση στην περίθαλψη, για την ψυχική υγεία για όλες τις γυναίκες. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδέσουμε ε, αυτό το ζήτημα ε, με την ε, κάκιστη κατάσταση που επικρατεί σε πολλά κράτη-μέλη και τα υποχρηματοδοτούμενα συστήματα ιατρικής ε, που φυσικά δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερα προσκόμματα για την πρόσβαση των γυναικών σε αυτές τις υπηρεσίες. Σίγουρα θα καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες, συνεργασία με τους συναδέλφους και με πεπισμένο θα είναι πάρα πολύ καλή η τελική έκθεση. Σας ευχαριστούμε. Κύριε δεν ξέρω μήπως έχει κάτι τόσο συμπληρωματικό να πει μετά από αυτά τα οποία είπαν και οι συνεισηγητές. Ένα σύντομο συμπέρασμα, λέει η κυρία Μπεθέρα, να υπενθυμίσω ότι έχουμε στην ουσία εδώ μπροστά μας, τα χέρια μας, ένα σημαντικό μέσο για να βοηθήσουμε να αλλάξει κάπως η κατάσταση κάνουμε μια κοινή διάγνωση ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι υπάρχει μια αντικειμενική ανισότητα στην πρόσβαση των γυναικών στην υγεία που είναι ένα αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Εδώ συμφωνούμε όλοι λοιπόν και θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω και μετά από τα σχόλια τα οποία έκανε η κυρία Πέτυρ ότι οι ιδεολογίες προφανώς και έχουν μια κάποια σημασία, σχετική όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ εκπροσωπούμε διαφορετικούς πολιτικούς προσανατολισμούς, διαφορετικές ιδεολογίες και πολιτικές ομάδες. Συμπίπτουμε όμως όλες λέγοντας ότι θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικές. Και είμαστε αποτελεσματικές πρώτον όταν έχουμε κάνει μια κοινή διάγνωση εντοπίζοντας τους τομείς τους οποίους τα πράγματα μπορούμε να τα βελτιώσουμε ή να διαπιστώσουμε και πού τα πράγματα πηγαίνουν καλά και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι τα αναγνωρισμένα δικαιώματα θα πρέπει να τα εφαρμόζουμε, να γίνονται σεβαστά και όλοι οι πολίτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αυτά. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό του πληθυσμού και δεν μπορεί να αποκλείονται γιατί τότε τα πράγματα δεν πρόκειται ποτέ να βελτιωθούν. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην κυρία Πετήρο ότι εγώ σε καμία περίπτωση δεν έχω α, κάποια, κάποιες ιδεολογικές προκαταλήψεις. Αυτό το οποίο όμως προσπαθώ και για το οποίο είμαι προκατηλημένη ουσιαστικά είναι η αποτελεσματικότητα. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικές εδώ, θα πρέπει να αποκλείσουμε κάθε τύπου α, κλισέ και εκ των προτέρων ιδεολειπτικές ε, απόψεις και να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας ε, στα πραγματικά θέματα, στα πραγματικά προβλήματα. Να αλλάξουμε λοιπόν έτσι τα πράγματα, ε, αυτή είναι η δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε, από κοινού θα πρέπει να την κάνουμε και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε τέτοιου είδους συμφωνίες οι οποίες ανεξάρτητα από κάποιες επιμέρους επιφυλάξεις και διαφωνίες θα βοηθήσουν να αλλάξουν τα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες λοιπόν για την προσπάθειά σας, για την δεκτικότητά σας, για την θετική σας στάση και νομίζω ότι και στα πλαίσια της συνάντησης των σκιωδών μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ε, μεγάλη εμβέλεια συμβιβαστικές τροπολογίες. Κυρία Μπεθέρα, να θυμίσω ότι είμαστε ένα όργανο πολιτικού χαρακτήρα ότι εδώ εκπροσωπούμε πολιτικές θέσεις, εκπροσωπούμε ιδεολογικές πολλές φορές θέσεις και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θα πρέπει να θεωρείται αρνητική η έκφραση μιας ιδεολογικής θέσης. Φυσικά δεν συμφωνούμε σε όλα τα θέματα Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις τις οποίες δεν συμμεριζόμαστε όλες αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ ακριβώς για να εκπροσωπήσουμε τη διαφορετικότητα των πολιτικών και ιδεολογικών μας θέσεων. Και μέσα από τις διαφοροποιήσεις αυτές τις πολιτικές και τις ιδεολογικές θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και να βρούμε ε, την σωστή λύση, τη συμφωνία. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε τις ιδεολογικές διαφορές, το πρόβλημα της ιδεολογίας σαν κάτι το αρνητικό. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα τώρα της ημερήσιας διάταξης. Έχει φτάσει πια η συγγήτρια της γνωμοδότησης ΣΥΝΚΟ για τη γυπνίαση των νομικών ρυθμίσεων και των διοικητικών μέτρων από πλευράς των κρατών μελών για την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Ε, Ευχαριστώ, αλλά ήμουνα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η ρύθμιση αυτή για την προσβασιμότητα προέρχεται από το άρθρο 9 της Σύμβασης των Μενωμένων Εθνών είχε υπάρξει το έτος αυτό προσβασιμότητας ήδη από το 2011 και εδώ και ένα χρόνο ενέκρινε τη συγκεκριμένη πράξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπήρξε και η απόφαση από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών πέρυσι το 2015 δηλαδή για το πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι ρυθμίσεις από τα κράτη-μέλη και είχε ζητηθεί να εγκριθεί η συγκεκριμένη αυτή νομική πράξη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν υπάρξει γνωμοδοτήσεις λοιπόν θετικές από πλευράς κοινοβουλευτικών επιτροπών. Υπάρχουν θετικές αντιλήψεις γύρω από τις προτάσεις αυτές, υπάρχουν όμως και κάποια πεδία βελτίωσης. Οι ρυθμίσεις αυτές θα είναι δεσμευτικές για τα κράτη-μέλη δεν απαιτούν ομοφωνία στο Συμβούλιο αλλά ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία απαιτείται σεβασμό συγκεκριμένων προδιαγραφών και υπηρεσιών όχι μόνο από τους κατασκευαστές αλλά και από τους διανομείς των προϊόντων από τους ε, εμπόρους ε, αυτούς οι οποίοι διοχετεύουν στις αγορές τα προϊόντα έτσι ώστε σε όλα τα προϊόντα παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων αυτών να παραμένουν διαθέσιμα, προσβάσιμα. Και υπάρχουν και συγκεκριμένες διαδικασίες λοιπόν για την προσβασιμότητα στα προϊόντα αυτά και τις υπηρεσίες. Υπάρχουν όμως και συγκεκριμένες προτάσεις επιμέρους βελτιώσεων είναι αν θέλετε περιφερειακές προτάσεις ε, γιατί όταν υπάρχει σαν παράδειγμα ένα προϊόν που δεν σέβεται την οδηγία αυτή να υπάρχει η δυνατότητα έτσι ώστε να μπορούν μετά από αιτήματα των οργανώσεων των καταναλωτών να υπάρξει σωστή ενημέρωση για τα προαπαιτούμενα της προσβασιμότητας να δημοσιεύονται τα προϊόντα αυτά και οι όροι μέσω των οποίων μπορεί να κυκλοφορήσουν, να δούμε ακριβώς τι γίνεται και με την πληροφορική, με τις νέες τεχνολογίες οι οποίες θα πρέπει να παραμένουν προσβάσιμες για όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν και για την εργασία, για τις κοινωνικές υπηρεσίες, για τις σπουδέ κτλ. Αυτές τις μέρες θα, δημιουργηθεί, θα συνέλθει το Ευρωπαϊκό Φόρουμ γύρω από τα θέματα αυτά και το οποίο θα συζητήσει πόσο μπορεί να, να συμπληρωθεί η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αφού έχουμε και την άποψη του φόρουμ αυτού θα καταθέσουμε την συνολική μας άποψη. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Η κυρία Χέντι. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ρώσα Φεραγκό, την εισηγήτριά μας, ε, για τη δουλειά που έχει κάνει. Φαίνεται ότι έχουμε επιτύχει μια προσέγγιση απόψεων για τα σημαντικότερα ζητήματα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό διότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η έκθεση. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εργαστεί σκληρά για την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις αγορές αυτές και υπάρχουν νέα απαιτήσει για τους οικονομικούς φορείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακολουθεί τη σωστή πορεία η πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να συμβάλλουμε και εμεί ούτως ώστε να ενισχύσουμε την τη θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενισχυμένη διαφάνεια για τις διαδικασίες καταγγελίας από πλευράς των καταναλωτών για τα προϊόντα ή για την παροχή υπηρεσιών, ε, συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, ε, με την αυξημένη διαφάνεια θα μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότερο στην ενιαία αγορά οι καταναλωτές ε, και οι οικονομικοί φορεί ε, θα συμμορφώνονται με τι υποχρεώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ο στόχο μα. Επίση, ε, οι οικονομικοί φορεί θα πρέπει να υπομιστούν ε, τι ευθύνε του ανεξάρτητα με το αν είναι παραγωγή, εισαγωγή ή διανομή δεν θα πρέπει να φέρουν το βάρος οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές ε, ευκολότερα θα πρέπει να ε, καταγγέλουν ε, αν χρειάζεται και να αναγνωρίζεται η ευθύνη των οικονομικών φορέων ώστε να αποφύγουμε και διακριτική μεταχείριση που πλήττει ε, τις γυναίκες και τα κορίτσια στον τομέα αυτό. Θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες. Προσβλέπουμε ανυπομονησία στη μελλοντική συζήτηση για την έκθεση και νομίζω ότι αν κρίνω από την πορεία της έκθεσης, θα, θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό κείμενο όπου θα φαίνονται οι προτεραιότητες που θέτει η Επιτροπή των Γυναικών. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κούνεβα, τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο οδηγία για την προσβασιμότητα σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίε είναι μια μεγάλη επιτυχία του κινήματο των ατόμων με αναπηρία. Φυσικά υπάρχουν πολλέ ελλείψει και όπω διαπιστώνει στη γνωμοδότηση τη συνάδελφο Εστάρα Φεραγκούτ, δεν είναι επαρκή οι απαιτήσει για το τοπιμένο περιβάλλον. Και είναι αλήθεια. Τα άτομα με αναπηρία στα περισσότερα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε είναι είτε αναγκάζονται να παραμείνουν αόρατα αφού με δυσκολία τολμούν να βγουν έξω από το σπίτι σε ένα περιβάλλον που δεν διαθέτει πρόσβαση στους δρόμους, στις πλατείες, στα πεζοδρόμια, στα νοσοκομεία, στα ιατρία και στα άλλα. Επίσης, συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά όχι μόνο στην προσβασιμότητα, αλλά και στις ίσες ευκαιρίες και τα δύο, και τα δύο φύλλα. Εδώ δεν είναι μόνο μια αναφορά. Το σχέδιο οδηγίας πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά και τις γυναίκες που είτε είναι σε εγκυμοσύνη, είτε έχουν το μωρό τους σε αμαξίδιο, είτε είναι προχωρημένης ηλικία. Επίσης, συμφωνούμε με την εισηγήτρια ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας μπορεί να διευρυνθεί ώστε να καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων. Για αυτό το λόγο, με τις τροπολογίες μας, θα προτείνουμε να γίνει επέκταση της προσβοσιμότητας σε οικιακές συσκευέ με διαποφή χρηστή, σε υπηρεσίε καλυμμάτων, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής διατυπώσης. Δικ, δικτύωσης. Επιπλέον, προσοχή πρέπει να δοτεί ιδιαίτερα στο κόστος. Τα άτομα με αναπηρία, τα οποία στην πλειοψηφία είναι χαμηλή στο εισοδομάτων δεν πρέπει να επιβαρυνθούν από το πιο κόστο των απαιτούμενων αναγκών. Τα νέα προϊόντα και υπηρεσίε πρέπει να είναι και οικονομικά προσβάσιμα. Τέλο, θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το κείμενο με δικλείδε ασφάλεια σε ό,τι αφορά πρώτο την ενίσχυση των υποπτικών αρχών. Δεύτερο, τις αναλυτικές επεξηγήσεις που τα συνδέονται τα νέα προϊόντα. Τρίτο, την κατάρτιση προσωπικού που θα βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιήσουν τα νέα προϊόντα. Τέταρτο, την γρηγορότερη εφαρμογή της οδηγίας στο χρόνο που προβλέπει η οδηγία, αφού ειδικά στα ηλεκτρονικά προϊόντα είναι πολύ μικρός ο χρόνος ζωής και τεχνολογικής ανανέωσής τους. Σε ευχαριστώ. Muchas gracias, señora Kuneva. Tiene la palabra la señora Reitke. Thanks a lot, Madam Chair, and thanks a lot to... Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για τη σύνταξη της γνωμοδότησης αυτής. Θα συμφωνήσω και εγώ με τους συναδέλφους. Έχουμε ήδη μια πάρα πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις. Και όλο αυτό αποτελεί κομμάτι ενός μεγαλύτερου πακέτου που αφορά την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Αθηνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Και οφείλω να ομολογήσω πως ε, η οδηγία είναι πάρα πολύ καλή, είναι νομικά δεσμευτική, αλλά αν δούμε το κείμενο, στο σύνολό του η εντύπωση που έχω αποκομίσει είναι ότι ε, λείπει η προσοχή στη διάσταση του φύλου. Και η Επιτροπή μας θα παίξει σημαντικό ρόλο εδώ, διότι όπως είπαν και οι συνάδελφοι, οι γυναίκες με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένες προκλήσεις και έχουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Γι' αυτό θεωρώ πως εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε αυτές οι συγκεκριμένες ανάγκες να καλύπτονται από τις δράσεις της Ένωσης στην προσπάθειά μας να ε, εφαρμόσουμε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, όπως αναφέρθηκε, οι γυναίκες δεν υποφέρουν από διακρίσεις όταν οι ίδιες πάσχουν από κάποια αναπηρία, αλλά ε, πολλές φορές φροντίζουν άτομα με αναπηρία και έχουν επιπτώσεις αυτές οι δράσεις και σε αυτές. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να καλύπτονται όλες οι πτυχές ε, του θέματος αυτού. Οι δικές μας τροπολογίες αφορούν την, παρά, την ε, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, να, έτσι ώστε να καλύπτει διάφορες δημόσιες πτυχές, να αφορά για παράδειγμα την προσβασιμότητα στο σπίτι, σε οικιακές συσκευές για παράδειγμα, και να φροντίσουμε όλο το νομοθετικό μας έργο να έχει μία εναρμονισμένη προσέγγιση για τα άτομα με αναπηρία και τις ανάγκες που υπάρχουν για περισσότερη προσβασιμότητα. Γι' αυτό λοιπόν να πω κλείνοντας πως μας χαροποιεί πολύ η πρόταση και ε, με χαρά θα συμμετέχουμε στην ανταλλαγή απόψεων. Η κυρία το Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω καταρχάς πως θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή της. Είναι μια ιδιαίτερα καλή γνωμοδότηση. Είναι μια γνωμοδότηση που ασχολείται με θέματα ουσίας. Τώρα να πω πως ε, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε για την οδηγία, ακόμα και εκτός αρμοδιότητας αυτής της Επιτροπής, ακούστηκε ότι η οδηγία αυτή είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και για το ευρύτερο κοινό. καθώς μεγαλώνουμε όλοι θα βρεθούμε σε μία θέση όπου θα αρρωστήσουμε ή θα ε, είμαστε προσωρινά ανίκανοι να εργαστούμε. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη για μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε όλους. Και αυτά ε, έδειξαν οι συζητήσεις με τους συναδέλφους. Πρέπει να δούμε όλες τις ε, πτυχές της οδηγίας, να τη δούμε σφαιρικά, γιατί είναι θέματα που μας αφορούν όλους. Θεωρώ επίσης ότι το σχέδιο γνωμοδότησης είναι κάτι αρκετά θετικό, διότι θα δώσει ευκαιρίες στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν νέους πελάτες, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Δεν πρέπει λοιπόν να περιοριστούμε στην προσβασιμότητα μόνο των υπηρεσιών, για παράδειγμα στην προσβασιμότητα σε ε, ε σε τράπεζες, σε τα σταθμούς. Πρέπει να δούμε το θέμα ε, σφαιρικά και να προσπαθήσουμε να εξελίψουμε τα εμπόδια προσβασιμότητας γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν μπορώ και εγώ να επαναλάβω αυτά που είπε η συγγήτρια, δηλαδή ότι χρειάζεται να συμπεριληφθούν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και διάφορε ενώσει που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία. Νομίζω πω ε, δεν υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Θα ήθελα όμω, εάν υπάρχει κάποιο, να ρωτήσω τι άποψη έχουν για το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η συγγήτρια. Προσωπικά θεωρώ πως ε, θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα συντομότερα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ίδια άποψη. Έχω και άλλες παρατηρήσεις, θα τις υποβάλω όμως γραπτός με τη μορφή τροπολογιών. Πάντως, κλείνοντας, θα ήθελα και εγώ να πω πως είναι ιδιαίτερα καλή η πρόταση της εισηγήτριας. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα ε, συγχαίρουμε την εισηγήτρια για την ποιοτική έκθεση και για την υποστήριξη που μας προσφέρει. Ευχαριστούμε και τους βουλευτές που τοποθετήθηκαν σχετικά και μας υποστηρίζουν ε, σε αυτή την προσπάθειά μας. Όντως είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπολογίζουμε στη βοήθειά σας για να το βελτιώσουμε. Κανένα κείμενο δεν είναι τέλειο. Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας για να βελτιώσουμε το κείμενο. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω κάποια επιμέρους σημεία. Προσπαθήσαμε κατά την εκπόνηση της θέσης μας να αποφύγουμε επιπρόσθετο διοικητικό άρθος ε, και για τη διοίκηση και για τις επιχειρήσεις. Κατανοούμε την επιθυμία σας για την ενίσχυση των ελέγχων, όμως ε, θέλαμε σε καθημερινή βάση να είναι διαχειρίσιμη η οδηγία για τις επιχειρήσεις που καλούνται να την εφαρμόσουν, αλλά και για την ε, δημόσια διοίκηση. Ευχαριστώ επίσης την προσοχή σας σε μια τροπολογία που σχετίζεται με το κείμενο στο τέλος του για τα άρθρα 27 και 28 της οδηγίας για ε, την ε, προθεσμία θέσης εφαρμογή και υποβολής αναφορών ζητάτε να επιταχυνθεί η διαδικασία και το καταλαβαίνουμε και φυσικά είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί το σχέδιο για την προσβασιμότητα σε σχέση με τι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει, τούτου λεχθέντω προσπαθήσαμε να είμαστε λογικοί ω προ τι προθεσμίε, κυρίω για του οικονομικού φορεί, ούτω ώστε να του επιτρέψουμε να προσαρμόσουν την αλυσίδα παραγωγής και άλλε πτυχέ για να συμμορφωθούν με τι υποχρεώσει, Δεν είναι πάντοτε προφανέ αυτό. Οπότε προσπαθήσαμε να βρούμε τη χρυσή τομή και να είμαστε και λογικοί για την προθεσμία για την υποβολή αναφορών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μείωση προθεσμία στα τρία χρόνια σας παραπέμπω στο άρθρο 28. Είναι ευρύτατο το πεδίο που θα καλύψει η αναφορά των πεπραγμένων και γι' αυτό και πρέπει να ε, ε, έχουμε υπαρκές πληροφορίες και να αναλύσουμε αυτές τις πληροφορίες που θα μας προσκομίσουν τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι πιο λογικό κάθε πενταετία να γίνονται οι ανταλλαγές, ούτως ώστε να είναι πλήρης η έκθεση προπραγμένων. Αν ε, σπέσουμε υπερβολικά, τότε ε, λόγια επικίνδυνο να μην είναι τόσο πλήρης η αναφορά όσο θα θέλαμε. Τέλος, ένα λεπτό. Α, ναι. Ε, υποστηρίζουμε τη γραμμή της εισηγήτριας η διαβούλευση θα πρέπει να έχει προτεραιότητα ε, με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ε, τα ΑΜΕΑ. Αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διαδικασία εφαρμογής οδηγίας και χαιρόμαστε που έχουμε και σε αυτό το σημείο την υποστήριξή σας. Ελπίζω να ήμουν αρκετά σύντομη και να έκανα ένα ικανοποιητικό απολογισμό της ε, το πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτήν την έκθεση. Ευχαριστούμε κυρία Σταρές για τα καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Υπήρχαν ορισμένες ανησυχίες για το αν όλες οι οργανώσεις αυτές οι οποίες είναι οι πιο έγκριτες θα έλεγα φωνές των ανθρώπων με αναπηρίες ε, να μπορούν να επηρεάσουν τη συζήτηση και να πάρουν μέρος στη συζήτηση. Τώρα για την εφαρμογή, την χρονική προθεσμία για την ε, εφαρμογή των προβλέψεων της οδηγίας να περάσουμε από τα 6 στα 5 χρόνια. Αυτό το είχε ήδη υποσχεθεί το 11 η Reading και το έκανε και το 12 και το 13 και το 14 και τώρα φτάσαμε και μετά το 2015. Συνεπώς λοιπόν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ε, αυτά τα οποία μας λέγουν. Σίγουρα ήταν ιδιαίτερα έντονη και οι προσπάθειες που έκανε η Επίτροπος για να περάσει η οδηγία αυτή. Ε, δυστυχώς τα χρόνια πέρασαν, τα πράγματα δεν έγιναν. Σίγουρα απαιτείται ένα χρονικό διάστημα και θυμάμαι μια οδηγία γιατί έγινε μια συζήτηση στην Γιούρη, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, η οποία λέει και στη συζήτηση φάνηκε ότι μια οδηγία για την ισότητα ανδρών γυναικών χρειάστηκε ε, λίγο πάνω από δύο χρόνια για να εφαρμοστεί. Συνεπώ τώρα να μιλάμε για έξι χρόνια είναι πάρα πολύ, είναι υπερβολικό. Νομίζω ότι τα πέντε χρόνια είναι αρκετό. Όταν βέβαια που να ξεκινήσει η διαδικασία είναι μια περίοδος η οποία προκαλεί μια κάποια αδράνεια, αλλά πάνω από πέντε χρόνια είναι λίγο υπερβολικό. Γιατί με τους αριθμούς παίζουμε πάρα πολύ εύκολα, είμαστε λίγο επιπόλαιοι θα έλεγα, ε, τι πέντε, τι έξι, τι εφτά ε, νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Ευχαριστώ την κυρία Εστάρας. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση είναι η 11η Νοεμβρίου στη μία το μεσημέρι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, 10 λεπτά. Θα διακόψουμε για 10 λεπτά. Ίσως να ξεκινήσουμε και λίγο μετά τις 5, αλλά στις 5 συνεδριάζουμε μαζί με την Επιτροπή Γεωργίας για την θέση της γυναίκας στην Ήπεθρο, στον αγροτικό χώρο. Λοιπόν, ένα γρήγορο καφέ, γιατί στις 5 και 5 ξεκινάμε.